Άρχεται η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση του κυρίου Κάμπρνοχ για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο ο εισηγητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σήμερα. Το θέμα μας είναι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφαλείας ε, στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου εδώ πέρα γιατί νομίζω πως μπορούμε να υπερψηφίσουμε την πρόταση αυτή με μια ευρεία πλειοψηφία. Στόχος του νέου κανονισμού είναι η μετανάστες από οποιοδήποτε κράτος μέλος, οι απάτριδες, οι πρόσφυγες να καλύπτονται ε, ανα πάσα στιγμή από συστήματα κοινωνικής ασφάλισης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Και να μην ε, λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα σε περισσότερες από μία χώρα. Η ερμηνεία λοιπόν της νομοθεσίας θα απλοποιηθεί. Υπάρχουν τρεις ε, βασικοί τομείς ε, εδώ πέρα. Έχουμε τον ε, ορισμό αρκετών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων εκτός του οικίου κράτους. Κατόπιν ορίζουμε ποια είναι η βάση ε, η έδρα στην ε, περίπτωση πληρωμάτων αεροσκαφών η οποία έδρα ή βάση τους ε, θεωρείται το αεροδρόμιο από το οποίο απογειώνονται και προσγειώνονται συχνότερα. Για να δούμε ακριβώς ποια νομοθεσία θα ισχύσει και μετά υπάρχει ο ορισμός του ανέργου και το τι σημαίνει αυτό. Κάποια κράτη-μέλη συμπεριλαμβάνουν και τους αυτοαπασχολούμενους στους άνεργους, άλλα κράτη-μέλη όχι. και αυτό καλύπτεται από την πρόταση κανονισμού. Δηλαδή, σύμφωνα με τον κανονισμό, ο αυτοαπασχολούμενος θα έχει τις καλύψεις του ανέργου στο κράτος μέλος το οποίο εργάστηκε για τελευταία φορά. Η αβεβαιότητα δε στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας επιλύθηκε και έτσι έχει επιληθεί το, το ζήτημα αυτό. Η με υψηλότερη προστασία η οποία παρέχεται σε μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων είναι οπωσδήποτε κάτι το θετικό για την ε, ενιαία αγορά. Και οι διατάξεις ε, περί ανεργίας οπωσδήποτε θα ωφελήσουν και τα άτομα εκείνα τα οποία θα καλύπτονται από αυτές. Σας ευχαριστώ. Επειδή ο Επίτροπος κάποιο πρόβλημα θα είχε και δεν παρίσταται, περνάμε στους ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων. Για δύο λεπτά, εξ ονόματος του ΕΛΚ, έχει το λόγο η κυρία Εσάγια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κρίμα που δεν μπόρεσε να έρθει ο Επίτροπος. Το Κοινοβούλιο παρακολούθησε τις εργασίες του Επιτροπής και του Συμβουλίου για το θέμα διότι στην ενιαία αγορά έχει κανείς το δικαίωμα να εργάζεται σε χώρα άλλη από την δική του. Παρόλα αυτά αυτό είναι μια πρόκληση. Δημιουργεί ορισμένα προβλήματα για τα κράτη-μέλη λόγω της διαφοράς των συστημάτων ασφάλισης και πρέπει να προβλεφθούν τρόποι καταπολέμησης των σχετικών απατών. Στόχος μας λοιπόν εδώ είναι να συντονιστούν τα συστήματα αυτά και να εξυγχρονιστούν λόγω των πρόσφατων αλλαγών. Να είναι σαφές τι ισχύει στην περίπτωση που κάποιος εργάζεται για σε χώρα άλλη από τη δική του. Βεβαίως δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό να αλλάζει συνέχεια ο ισχύων νόμος επειδή κάποιος αλλάζει χώρα εργασίας. Πρέπει να ισχύουν τα ίδια παντού. κάποιος άνεργος αυτοαπασχολούμενος πρέπει να μπορεί να επωφελείται από τα επιδόματα ανεργίας στη χώρα στην οποία εργαζόταν. Ακόμη και αν δεν προβλέπεται τέτοιο επίδομα στη χώρα διαμονής του. Η πρόταση έχει προσαρμοστεί για να εφαρμόζεται μόνο σε καθαρές περιπτώσεις τέτοιων διαμεθοριακώς εργαζομένων. Και σε δύο χρόνια προβλέπεται να αναθεωρηθεί για να δούμε αν προκύψει κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Εσαγιά. Έχουμε τώρα τον Επίτροπο. Γι' αυτό θα του δώσω το λογορίστε κύριε Επίτροπέ μου. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητά ε, μέλη. Το θέμα συζήτησης ορίζει ειδικά μέτρα για τον συντονισμό των εθνικών συστημάτων ασφάλισης για να ε, μπορέσουμε να υπερασπίσουμε τους απασχολούμενους που εργάζονται διασυνοριακά. Γι' αυτό θα πρέπει να αντικαταπτρίζουν την νομική και κοινωνική κατάσταση. μετά από, τον, από την αναθεώρηση τον κανονισμών το 2010 είδαμε ότι υπάρχουν αλλαγές στην εθνική νομοθεσία και, και γι' αυτό επειδή πρέπει να επέλθουν ακόμα περισσότερες η πρόταση που συζητεί σήμερα το Κοινοβούλιο, που συζητά σήμερα το Κοινοβούλιο, λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις που δεν είχαν ληφθεί υπόψη εν λεπτομερία στον κανονισμό. Ε, είναι βεβαίως τεχνικής φύσης ο κανονισμός, έχει όμως επιπτώσεις στους εργαζόμενους όταν χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης. Με βάση το ε, ψήφισμα και την έκθεση του 2010 τονίζουμε ότι η ελεύθερη διακίνηση θα πρέπει να δίνει, να συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα, ιδιαίτερα ως προς την εγκατάσταση και αφορά τα δύο πιο ευαίσθητα ζητήματα, την αρχή της διαμονής για τα πληρώματα και τα επιδόματα ανεργίας για τους αυταπασχολούμενους που επιστρέφουν στην χώρα διαμονής αλλά όπου δεν υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα, δεν προβλέπεται. Ο συμβιβασμός στον οποίο φτάσαμε συνοδεύει το πνεύμα του κανονισμού, συνάδει με το πνεύμα του κανονισμού ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων και όταν ε, εφαρμόζεται αυτό το νομικού περιεχομένου κείμενο. Ο κύριος Καμπρνόχ θεώρησε ότι θα πρέπει να εγκριθεί το θέμα σε πρώτη ανάγνωση μετά από τις περισσινές διαπραγματεύσεις και είμαι ευγνώμων διότι έλαβε υπόψη τις δικές μας θέσεις στα ψηφίσματα συμβασμού, έτσι ώστε να προωθηθεί η συνεργασία των δύο θεσμικών οργάνων σε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε κύριε πίτροπε. Το λόγο έχει εξ ονόματος των σοσιαλιστών και δημοκρατών ο κύριος Θέρκας για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κάμπρνοχ αλλά και την Επιτροπή για την εξαιρετική εργασία γιατί βρήκαμε έναν τρόπο επίλυσης του θέματος με την αναδιατύπωση και επικαιροποίηση αυτού του κειμένου για τους δικαιούχους, για τους άμεσους δικαιούχους. Νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό εάν λάβουμε υπόψη τα επιδόματα ανεργίας για τους ε, διακινούμενους εργαζόμενους και αυτό θα ισχύσει σε δύο χρόνια για να μπορέσουμε να ε, επιλύσουμε και το θέμα του άρθρου 11 για τα πληρώματα ε, αεροσκαφών, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη την έννοια του home basis, την έδρα βάσης. Σήμερα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πώς η Ευρώπη μπορεί να βελτιώσει την εργασία χιλιάδων εργαζομένων μέσα στα πλαίσια καταστάσεων υψηλής ανεργίας και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβάλλει πρότυπα αντιμετώπισης της ανεργίας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση διότι αυτό ζητάει η κοινωνική ατζέντα και μπορούμε να το καταφέρουμε σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Θέρκας. Information Μία πληροφορία για, για, τους, ε, ε, για τον εισηγητή. Ε, νομίζω ότι το όνομά του προφέρεται Σάρνοχ. Και αυτό το λέω για τους υπόλοιπους, για, ιδιαίτερα για τους κατοίκους Μεσογείου που δεν μπορούν να προφέρουν εύκολα τσεχικά ονόματα. Η κυρία Οβίρ, εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Το δικαίωμα να δουλεύει και να εργάζεται κανείς σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης είναι δικαίωμα όλων των πολιτών της ε, Ένωσης. Εξάλλου η κινητικότητα της εργασίας είναι βασικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πυλώνας ε, της ενιαίας αγοράς και απαιτεί άρα συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Δεν θα πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος για τα της ανεργίας, της υγείας, της σύνταξης και τα λοιπά ζητήματα της ε, κοινωνικής ασφάλισης. Ο κανονισμός ο υφιστάμενος ε, είναι 10 ετών, η αγορά εργασίας έχει αλλάξει εντελώς, υπάρχουν νέες μορφές μετανάστευσης, γι' αυτό χρειάζεται και η επικαιροποίηση του κανονισμού. Η δικιά μας δουλειά ως κοινοβούλιο είναι να φροντίσουμε το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης σύμφωνα με το άρθρο 48 της συνθήκης να είναι εγγυημένο κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ε, των κοινωνικών εταίρων. Έχουμε τον ορισμό της ε, βάσης, ε, της έδρας των πληρωμάτων αεροσκαφών. Αυτά δεν απαιτούν από τα κρατημέλη αλλαγή της νομοθεσίας. Οι αλλαγές στον κανονισμό είναι προς το συμφέρον των πολιτών των 27 κρατών μελών και θα ισχύσουν και σε Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία. Το σκεπτικό εδώ πέρα είναι να αντικατασταθούν οι διμερείς συμφωνίες με ένα ενίο καθεστώς για να πληρώνονται πιο γρήγορα οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Σάμπερνοχ ε, και τους και για την γρήγορη και ποιοτική δουλειά τους. Σας ευχαριστώ κυρία Οβίρ. Το λόγο έχει για τους πράσινους ε, για δυόμιση λεπτά η κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι πράγματι τεχνικό το έγγραφο και πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως υπόθηκε. Αυτό το οποίο έχουμε εδώ πέρα είναι μια επικαιροποίηση της παλαιότερης ίσως ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έχαμε την αναθεώρηση που τελείωσε το 2009 και έχουμε τώρα την επικαιροποίηση. Σύντομα νομίζω θα δούμε το πώς ε, θα λειτουργήσει το νέο ηλεκτρονικό σύστημα και που ελπίζουμε να είναι γρηγορότερο στην αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών. Γιατί μιλάμε για την διατήρηση δικαιωμάτων ανθρώπων που έχουν διασχίσει σύνορα για οποιοδήποτε λόγο, είτε εργάζονται σε μυθεριωκές περιοχές, είτε όχι, για παροχή υγείας, ε, επιδομάτων ανεργίας κτλ και βέβαια πρέπει να υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα. Αυτό το οποίο έχουμε εδώ πέρα είναι ένα αποτέλεσμα φιλικό προς τους πολίτες ε, στη συμφωνία αυτή η οποία είναι στην πρώτη ανάγνωση. Όπως υπόθηκε, στόχο έχει να διατηρήσει τα δικαιώματα των ατόμων που καλύπτονται από κοινωνική ασφάλιση. Δεν ε, δημιουργήθηκε ε, για να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων και να δοθεί ε, ευκαιρία σε όσους έχουν ε, μετακινούμενους εργαζόμενους να επιλέξουν το φτηνότερο τρόπο ε, και τόπο εγκατάστασης. Χαίρομαι λοιπόν που καταφέρουμε να κλείσουμε το παραθυράκι αυτό. Γιατί το να βρεθεί κανείς εγγεγραμμένος σε μια χώρα με την οποία θεωρεί πως δεν έχει σχέση και να αναζητήσει υπηρεσίες υγεία στη χώρα στην οποία κατοικεί θα δημιουργήσει οπωσδήποτε προβλήματα για το άτομο αυτό παρά το ότι βεβαίω η εταιρεία θεωρεί πως ε, κερδίζει. Δεν είναι δίκαιο αυτό για τους ε, εργαζόμενους. Χαιρόμαστε λοιπόν τώρα για το ότι μπήκε εδώ πέρα ο ορισμός ε, περί βάσεις, αεροδρομίου για να ξέρουν και οι εργαζόμενοι τι δικαιώματα θα έχουν. Πολύ θετικό αποτέλεσμα λοιπόν και χαιρόμαστε που πέρασε στην πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστούμε κύριε Λάμπερτ. Εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών έχει το λόγο κυρία Γιανακουδάκη. Ευχαριστώ. Σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διευκολύνει τις επιχειρήσεις. Ως πρώην επιχειρηματίας ξέρω ότι είναι λογικό για τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος, τις δαπάνες τους. Όμως δεν θα πρέπει να υπεκφύγουν των υποχρεώσεων να καταβάλουν κοινωνική ασφάλιση. Το Λονδίνο, ε, η εκλογική μου περιφέρεια, είναι ο μεγαλύτερος επενδυτικός ε, χώρος και κόσμος. Όταν λοιπόν οι επενδύσεις όπως η Microsoft και η Sony επενδύουν στο Λονδίνο θα πρέπει να ενταχθούν στο Βρετανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Το ίδιο αφορά για εργαζόμενους που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώς ένα παραθυράκι ε, επέτρεψε στα πληρώματα στις αεροπορικές εταιρείες να μην ακολουθήσουν αυτό το πρότυπο. Δηλαδή, ορισμένοι εργαζόμενοι του Βελγίου που εργάζονται στην Ιρλανδία ή στην, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, καταβάλουν την κοινωνική ασφάλιση εκεί όπου έχει νιολογηθεί το αεροσκάφος, δηλαδή στην Ιρλανδία άρα δεν καταβάλουν κοινωνική ασφάλιση στην έδρα τους. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί έκλεισε αυτό το παραθυράκι και έτσι ε, μπορούν τα, τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης να έχουν τα έσοδα που χρειάζονται. Ευχαριστούμε κυρία Γιανακουδάκη εξ ονόματος της Ομάδας Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Το λόγο έχει ο κύριος Σιμάνσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση που συζητάμε αφορά το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Θέλουμε ίση μεταχείριση των πολιτών στην αγορά εργασίας και γι' αυτόν τον λόγο οι αλλαγές στο κα... ισχύοντες κανόνες πρέπει να προωθούν την κινητικότητα ιδίως των ανέργων. Δεν πρέπει τεχνητά να αναγκάζεται κανείς να διαμένει εκεί που εργάζεται απλώ και μόνο γιατί μόνο εκεί του χορηγούνται δικαιώματα. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την έκθεση. Καλύτερο συντονισμός των συστημάτων ε, κοινωνικής ασφάλισης θα ήταν ένας τρόπος για να διασφαλίσουμε μια εξισορρόπηση μεταξύ ανταγωνιστικότητας και προστασίας των εργαζομένων. Η πρωτοβουλία του Κομισιόν του περασμένου Μαρτίου για τους προσωρινώς αποσπασμένους αφορούσε ένα εκατομμύριο εργαζόμενους και είναι σχετική με αυτό το πρόβλημα που συζητάμε. Η ανταγωνιστικότητα και η προστασία των εργαζομένων είναι δύσκολο να εξισορροπηθούν αλλά είναι απαραίτητο σε αυτή την εποχή που ζούμε τέτοια κρίση. Ευχαριστούμε κύριε Σιμάνσκι. Τώρα η κυρία Ζούμπερ. Θεωρούμε ότι ένας αυτοαπασχολούμενος που μισθοδοτείται θα πρέπει να καταβάλει ε, και την κοινωνική ασφάλιση στο κράτος που εργάζεται. Θεωρούμε όμως ότι η έννοια της ε, βάσης έδρας είναι πολύ σωστή. Όμως αυτό το μέτρο δεν θα πρέπει να νομιμοποιήσει τους απασχολούμενους, δηλαδή εκείνους που απασχολούν μία θέση αορίστου χρόνου. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε συμβάσεις αορίστου χρόνου, οι οποίες να διέπονται από μία διαφορετική ε, βάση επίσης. Ως προς τα πληρώματα θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος στην έδρα βάση έτσι ώστε να μην υπάρχει υπεκφυγή και καταβάλλονται τα επιδόματα σε χώρα με χαμηλότερο κόστος. Τη στιγμή που υπάρχει, γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος κατά του εθνικού μας συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, δεν θα δεχτούμε το ευρωπαϊκό σύστημα συστάσεων που στην ουσία επιβάλλονται, όπως τη Λευκή Βίβλο συνταξιοδοτήσεων ή ιδιωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να μην δεχτούμε τις περικοπές που γίνονται και στις αδειοδοτήσεις και στα κοινωνικά επιδόματα. Εμείς είμαστε υπέρ ενός ε, δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την καθολικότητα δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε την κυρία Ζούμπερ. Εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων, η κυρία Βέρμεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο νέος κανονισμός ε, δημιουργεί σαφήνεια για όλους τους ενδιαφερόμενους, ασφαλιστικά ταμεία, τους πολίτες και τις εταιρείες. Ε, ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως λαμβάνει υπόψη την κατάσταση ανθρώπων με μεγάλη κινητικότητα. Κάτι το οποίο χρειαζόμαστε είναι δίκαιη κοινωνικά, δεν έχει επιπλέον κόστος και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στους πολίτες. Ιδιαίτερα σημαντικές μου φαίνονται δύο πτυχές. Πρώτον, ή ε, ο σαφής καθορισμός ε, του όρου ουσιαστικό ποσοστό της εργασίας και δεύτερον ο ορισμός ε, της βάσης από την οποία ξεκινούν τα πληρώματα αεροσκαφών. Έτσι υπάρχει σαφήνεια πλέον για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και δεν υπάρχει κοινωνικό dumping. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα σε, στους άλλους ομιλητές. Ο κύριος Έρη έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πολλά ακούστηκαν ήδη στην συζήτηση. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Θα ήθελα όμως ε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία εμείς οι βουλευτές ε, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος ε, σε αυτά τα οποία απασχολούν τους ε, πολίτες. Αν θέλουμε να αποδείξουμε τη χρησιμότητα της δουλειάς της δικιάς μας και της Κομισιόν, αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει. Θεωρώ λοιπόν πως μέσω της ε, καλής και λογικής συνεργασίας μπορούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες να, έχουν, ε, να προσφέρουν διασυνοριακές υπηρεσίες και να συνεχίσουν να έχουν τις κοινωνικές τους παροχές. Ιδιαίτερο πλεονέκτημα της ε, συζήτησης αυτής και του συντονισμού είναι πως ε, βασιζόμαστε εδώ πέρα στις προτάσεις της Κομισιόν, τις εμπειρίες των ε, κρατών μελών και προσπαθούμε να απαντήσουμε τα τεχνικά ερωτήματα ήδη στην πρώτη ανάγνωση. Υπάρχουν πολλά μοντέλα απασχόλησης που είναι καινούρια υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο κινητικοί από ό,τι στο παρελθόν όσον αφορά την απασχόληση. Γι' αυτό χρειάζεται ε, μια προσαρμογή του νομικού πλαισίου για να υπάρχει μια ενιαία νομική αντιμετώπιση και θεωρώ πως ε, προσφέρουμε εδώ πέρα ένα πολύ καλό παράδειγμα αν είναι να έχουμε νέα μοντέλα και νέες λύσεις, τότε νομίζω πως είναι δημιουργική η λύση ε, που δώσαμε για τα πληρώματα των αεροσκαφών και θέλω άρα να σας ευχαριστήσω και εγώ ελπίζω η λύση την οποία βρήκαμε και θα μας απασχολήσει νομίζω το ζήτημα αυτού συντονισμού. Η κυρία Στάινουρκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή και χαιρετίζω την έκθεση αυτή. Η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά έχει πολλά πλέον εκτίματα, αλλά υπάρχουν κενά στην νομοθεσία τα οποία εκμεταλλεύονταν οι εταιρείε και αναφέρθηκαν διάφορα παραδείγματα όπως οι αεροπορικές εταιρείε. Συχνά κανόνιζαν τα δρομολόγια έτσι ώστε να ασφαλίζονται τα πληρώματα στο φτηνότερο κράτος. Και έτσι υπήρχε και στρέβλωση του ανταγωνισμού και υπήρχε κοινωνικό ντάμπινγκ. Γι' αυτό εμείς ως Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες θελήσαμε να καλυφθεί και το προσωπικό των ε, αεροσκαφών εκεί όπου έχει την βάση του. οι εργοδότες οι οποίοι εκμεταλλεύονται μόνο την εσωτερική αγορά χωρίς να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δεν έχουν θέση στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαρνέσκι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε από έναν ε, συνάδελφο, από ένα μέλος που ανήκει στην ίδια πολιτική ομάδα με μένα. Και τον υποστηρίζω όχι μόνο επειδή ανήκουμε στην ίδια ομάδα, αλλά επειδή πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική. Εδώ ακολουθούμε ένα είδος ε, όρκου του Ιπποκράτη. Δεν θα πρέπει να βλάψουμε ούτε τους εργαζόμενους αλλά ούτε τις επιχειρήσεις. Ούτε. Σε μία ε, οικονομική κρίση δεν θα πρέπει να βλάψουμε υπερβολικά ούτε τον ένα ούτε τον άλλο τομέα. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσαρνάτσκι. Ο κύριος Πάσκα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ένας από τους βασικούς όρους για την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων αφορά το εξής, τον συντονισμό των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κανονισμός 987 ε, του 2009 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, μάλλον να επικαιροποιηθεί. Και ο ορισμός Ο κανονισμός 883 του 2004, άρθρο 3, παράγραφος 1, είναι ύψης της σημασίας, δηλαδή η ερμηνεία για τους πολίτες μας, να υπάρχει καλύτερη προστασία για τους αυτοαπασχολούμενους, ιδιαίτερα όταν καθίστανται άνεργοι. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει και να δούμε βεβαίως εάν υπάρχει και πιθανότητα απάτης. Ο κύριος Όμπερμαϊερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης υπάρχουν νέες μορφές κινητικότητας, ε, όπως π.χ. τα πληρώματα αεροσκαφών και δεν θα πρέπει βεβαίως ε, να υφίστανται οι άνθρωποι αυτοί οι αρνητικές διακρίσεις. Αλλά δεν θα πρέπει να ε, επηρεαστεί η παροχή ε, κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα πρέπει να ε, υπάρξει παροχή κοινωνικών επιδομάτων σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι φορείς αυτών των δικαιωμάτων, όπως είχαμε πρόσφατα μία περίπτωση στην Αυστρία για Γάλλους υπηκόους οι οποίοι ζήτησαν ε, αυστριακά κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τουρισμό κοινωνικών παροχών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εάν είναι να λειτουργεί σωστά η εσωτερική αγορά, θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη ε, διακίνηση των εργαζομένων και παροχή ε, των ε, κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν αλλάζουν κράτη. Με τις νέες αυτές διατάξεις δεν, πρέπει κανείς να, δεν θα μπορεί κανείς να απορρίψει μία προσφορά εργασίας γιατί δεν θα ξέρει θα, ποια θα είναι τα δικαιώματά του. Επίσης αλλάζουν τα δικαιώματα για όσους δουλεύουν σε μεθοριακές ζώνες. Εκεί όπου εργάζεται θα έχει και κοινωνική προστασία κανείς. Αν όμως δουλεύει κανείς 25% του χρόνου στον, στη χώρα κατοικίας του, εκεί θα έχει και προστασία ε, ανεργίας. Επίσης βελτιώθηκε η κατάσταση για τα πληρώματα των αεροσκαφών για να μην διαλέγουν οι εταιρείε την έδρα τους κατά το δοκούν. Έχουμε επίσης αφαιστερούς ε, κανόνες και θα έχουμε αργότερα φέτος για τους αποσπασμένους. Ευχαριστούμε κύριε Κρίστενσεν. Περνάμε στο Catch the Eye. Ο κύριος ε, Νικολάτσης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία. συνεργάστηκε με όλες τις πολιτικές ομάδες που είναι σημαντικό πράγμα διότι ο κανονισμός αυτός ενδιαφέρει πολλούς στην Ευρώπη που θέλουν να επωφεληθούν από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Είναι κάτι που ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα τους εκλογείς μας. Η διαμεθοριακή εργασία είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό δεν είναι μόνο εκείνοι που εργάζονται σε άλλη χώρα από την χώρα προέλευσής τους. Υπάρχουν και εκείνοι που, που λέγω, που εργάζονται στις αεροπορικές εταιρείες. Πρέπει να ξέρουμε πώς πληρώνονται οι κοινωνικές παροχές σε τέτοιες περιπτώσεις με όση διαφάνεια χρειάζεται. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό η κυρία Ζαζοβιέτκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η νομοθεσία των μελών έχει... Η νομοθεσία χωρών μελών τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αλλάξει πολύ καθώς και η συμπεριφορά των ανθρώπων εργάζονται σε άλλες χώρες, υπάρχουν εταιρείε που η οικονομική τους δραστηριότητα ε, ασκείται σε διάφορες χώρες και οι αλλαγές αυτές δεν προκύπτουν μόνο από την κρίση αλλά από τις αλλαγές γενικότερα στην αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν να εξυγχρονιστούν οι κανόνες έτσι ώστε η κινητικότητα των εργαζομένων και η δυνατότητα των εργοδοτών να ασκούν την εργασία τους να διευκολύνεται. Οι αλλαγές λοιπόν της νομοθεσίας των χωρών μελών ως ανταπόκριση στην κρίση πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την αύξηση της κινητικότητας και αυτό απαιτεί περαιτέρω αλλαγές στα επόμενα χρόνια. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να σκεφτούμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και ένα μεγαλύτερο συντονισμό στα συστήματα κοινωνικής περίθαλψης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ζαζοβιέτκα. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Τζίνκιμπιτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή, ειδικά στο κομμάτι που αφορά τις αλλαγές μεταξύ συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εγώ είμαι υπέρ των ε, αλλαγών ε, που ενισχύουν την κινητικότητα των πολιτών. Η κατάσταση ενός αυτοαπασχολούμενου ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα κράτος μέλος και έχει δικαιώματα παροχών και μετά πηγαίνει σε άλλη χώρα όπου χάνει αυτά τα δικαιώματα δεν είναι αποδεκτή σε μια ε, Ευρώπη. Το ΔΕΚ ε, επίσης επιβεβαίωσε πως ε, τα άτομα τα οποία εργάζονται σε άλλη χώρα από τη χώρα την αρχική δικαιούνται και εκεί πέρα τις κοινωνικές τους παροχές ιδιαίτερα όταν η παροχές αυτές ε, συνδέονται με την εργασία τους. Σας ευχαριστώ κυρία Μπασέσκου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποστηρίζω και εγώ τον, την τροποποίηση των κανονισμών για τη συντονισμό και τη θέση εφαρμογή των συστήματων κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι θα βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου. Λαμβάνουμε υπόψη τις αλλαγές των εθνικών νομοθεσιών καθώς και τις ε, πλέον ε, πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της διασυνοριακής ε, διακίνησης. Έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε την εργατική δύναμη ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι πλήττονται πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους εργαζόμενους διότι υπάρχουν περισσότερα προαπαιτούμενα σε μία αγορά εργασίας που είναι υπερανταγωνιστική. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των πολιτών μέσω των επιδομάτων ανεργίας. Άρα υποστηρίζω την τροποποίηση του άρθρου 65 έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις ε, ε, διατάξεις στο νομοθετικό πλαίσιο με βάση την κοινωνική κατάσταση. Ο κύριος Μπάτεν έχει το λόγο για ένα λεπτό. E Μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης ε, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν σημαίνει θα ε, εναρμονίσουμε και τα συστήματα κοινωνικών επιδομάτων, αλλά την εναρμόνιση πρόσβασης σε αυτά τα συστήματα από όλους τους ε, πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί ε, θα προβάλλουν αξιώσεις στα γενναιόδερα συστήματά μας. Έχουμε 5 εκατομμύρια ετούντες και δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα συστήματα ε, στέγασης, στη χορήγηση στέγης. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν καταβάλει ναι, ναι, ναι. τίποτα καθόλου ε, στην κοινωνική ασφάλιση και παράλληλα θα στεγάζονται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο τα ε, ευεργετήματα αυτά είναι ή δεν είναι ε, αμοιβαία. Κανένας δεν, μπορεί, δεν θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει αυτά τα επιδόματα στέγασης ή ανεργίας εάν δεν έχει καταβάλει κοινωνική ασφάλιση στο ενομένο Βασίλειο. Λούμαν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, δέχομαι την βελτίωση αυτού του κανονισμού. Όπως ξέρετε, από την αρχή της θητείας θεώρησα ότι θα πρέπει να απλουστευτεί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να λειτουργεί καλύτερα και να ανταποκρίνει τις ανάγκες των πολιτών. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα θετικό βήμα ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και για την εμφάνιση της διακίνησης των εργαζομένων. Οι δύο κανονισμοί και ιδιαίτερα 883 του 2004 βελτιώνει την κατάσταση. Πέρα από αυτές λοιπόν τις ε, προαπαιτήσεις θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν τη σωστή εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έτσι ώστε αυτοί οι κανονισμοί να ε, ισχύουν σωστά για όσους εργάζονται ή πάβουν να εργάζονται σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Φλασίκοβα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ο στόχος ε, του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης έχει στόχο να συγχρονίσει το κεκτημένο. Η κοινωνία αλλάζει και άρα προτείνουμε και εμείς αλλαγές στην νομοθεσία περί ανεργίας. Στην περίπτωση που κάποιος εργάζεται σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη, ο ορισμός του σημαντικότερου τμήματος των δραστηριοτήτων τους ισχύει επίσης για ανθρώπους που έχουν πάνω από έναν εργοδότες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση ατόμων με πολύ υψηλή κινητικότητα. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν ε, κοινωνικά επιδόματα σύμφωνα με την ε, νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους και να έχουν την δυνατότητα βεβαίω να δουλέψουν όπου εγκατασταθούν. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριος Μπρόνους. Ό,τι και να συζητάμε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, δηλαδή περαιτέρω οικονομική και πολιτική ενοποίηση. Παλαιά, επί ΕΟΚ, μας έλεγαν πως είχαμε το δικαίωμα να εργαστούμε σε άλλες χώρες. Εάν δεν υπήρχε δουλειά, επέστρεπε κανείς στη χώρα του. Τώρα έχουμε ελευθερία διακίνησης των ανθρώπων που ζητάνε επιδόματα. Εδώ πέρα το παρουσιάζεται ως δίχτυ προστασίας ε, εργαζομένων που έχουν δυσκολίες, ενώ κίνητρο είναι να στηριχθεί ένας πολιτικός στόχος η μεγιστοποίηση της κίνησης των ανθρώπων για να υποβαθμιστεί η εθνική ταυτότητα. Σύμφωνα με τα λόγια του εισηγητή, θα υπάρξει χωρίς αυτό το συντονισμό η δυνατότητα να μην υπάρξει ε, ε, ελευθερία διακίνησης. Στόχος εδώ πέρα δεν είναι να ικανοποιηθεί κάποια ανάγκη των αυτοαπασχολούμενων, είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για να δημιουργηθεί ακριβώς αυτή η ζήτηση. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος. Ε, ε, Νομίζω ότι βασιζόμαστε στην προϋπάρχουσα νομοθεσία έτσι ώστε οι πολίτες να είναι δικαιούχοι κοινωνικής ασφάλισης όταν, όταν ε, μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο. Θα πρέπει όμως να βρούμε έμπρακτες λύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτό αφορά και την απόσπαση των εργαζομένων και την σχετική οδηγία, η οποία μας βοήθησε βεβαίως. Υπάρχουν επιπτώσεις και στο θέμα στέγασης ή έλλειψης στέγησης και σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Η πρόταση που συζητήθηκε μιλά για τεχνικές προϋποθέσεις για το συντονισμό στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης έτσι ώστε ο συντονισμός να αποτελέσει πραγματικότητα για τους πολίτες. Η Επιτροπή προσβλέπει στην έγκριση της πρότασης κατά την πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχει το λόγο, ε, έχει το λόγο εσύ της ο κύριος Σάμπρνοχ. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα εντάχει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την υποστήριξη και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Όπως ε, ακούσατε, όλοι τάσσονται υπέρ των αλλαγών αυτών που δεν είναι τεχνικής υφής αλλά και πολιτικής πρόταση αυτή υποστηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου πολιτών αυτοαπασχολουμένων, απλουστεύει τα πράγματα, τα καθιστά πιο απλά και σαφή γιατί μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο για τον ε, επιχειρηματικό κόσμο. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε με γραφειοκρατία τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να πω ότι η δυνάμη των προτάσεων αυτών τα προνόμια των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης ε, την χάνουν εγγυήσεων και δεν έχουμε ε, απαράδεκτες προσδοκίες. Μιλάμε για καθήκοντα και δικαιώματα των εργαζομένων μέσα στα πλαίσια μιας εξισορρόπησης. Άρα μιλάμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως θα πρέπει να λειτουργεί. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Η κυρία Τσασλοβιέσκα ζητάει το λόγο. Θα ήθελα για το επόμενο θέμα να λάβω το λόγο. Α, μάλιστα. Α, καλά. Φοβερό πράγμα. Βεβαίως να προετοιμάζεστε για το μέλλον. Το σημειώσαμε. Pues, eh, Κλείνει η συζήτηση επί του θέματος αυτού. Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στις 11.30. Ε, και τώρα διακόπτουμε για λίγα λεπτά μέχρι τις 10. Διακόπτουμε για λίγα λεπτά, για 2-3 λεπτά.